για την ασφαλή χρήση των ε, συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών RPAS στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Ελπίζω να γίνει λίγη ησυχία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Τα μικρά τηλεκατευθυνόμενα ε, χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1935 που είχε χρησιμοποιήσει και το Βρετανικό Ναυτικό ένα τέτοιο σύστημα. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αύξηση της χρήσης ε, ε, των drone όπως λέγεται, των τηλεκατευθυνωμένων ή τηλεχειριζομένων αυτών μηχανισμών και για εμπορικούς λόγους. Πρέπει να τεθούν λοιπόν τεχνολογικά όρια όπως επίσης και διακανονιστικά όρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα πολιτικής αεροπορίας όπως το Horizon 2020 και το Caesar. Είναι κάτι που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουμε υψηλά επίπεδα και στην κατασκευή των συγκεκριμένων μηχανισμών. 2.500 ε, χρήστες υπάρχουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάνω από 600 τέτοιες υπηρεσίες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όπως αεροφωτογραφίες κτλ. Ε, αντικαθιστούν τη χρήση αεροσκαφών για τέτοιου είδους φωτογραφίσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη σχεδίαση και τον έλεγχο σιδηροδρομικών γραμμών, ε, αθλητικών σταδίων, χρησιμοποιούνται επίσης και στην καταπολέμηση πυρκαγιών και στην προσπάθεια διάσωσης πολιτών που έχουν χτυπηθεί από σεισμούς κτλ. Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα baby drones που είναι και αυτά ιδιαίτερα δημοφιλή για λόγους ε, διασκέδασης. Ε, πρέπει λοιπόν, αν υπάρξει ένα πλαίσιο διακανονιστικό, να επιτρέπει την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής και εγώ σαν εισηγήτρια προσπάθησα να βρω το σωστό πλαίσιο έτσι ώστε η βιομηχανία αυτή να περάσει στην επόμενη φάση. Η έκθεση αυτή ως έχει δίδει απαντήσεις στις κεντρικές ερωτήσεις οι οποίες τίθενται. Εγώ συναντήθηκα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των κρατών μελών, των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας Αερομεταφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι αναγνώρισαν ότι όποιο πλαίσιο προταθεί θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες και στην αξιολόγηση κινδύνου έτσι ώστε να αποτραπούν αδικαιολόγητα εμπόδια. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή συνεργασία επίσης η οποία θα τονώσει και την έρευνα και την ανάπτυξη. Συναντήθηκα στη Ουάσιγκτον τον Μάρτιο και με εκπροσώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ε, και στην συνάντηση υψηλού επίπεδου ε, στη Ρήγα ε, τέθηκε το θέμα αυτό ελέγχθη ότι η κοινότητα των πολιτικών αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει από το 2016 με νέα μέτρα τέτοιου είδους δραστηριότητες. Απαιτούνται να υπάρξουν ευρωπαϊκοί και σφαιρικοί θα έλεγα παγκόσμιοι κανόνες και στον τομέα της αδειοδότησης, της εμπορικής χρήσης, της πιστοποίησης. Ε, όπως επίσης της προστασίας της ιδιωτικότητας και του καθορισμού των ε, περιοχών στις οποίες απαγορεύεται κάθε φορά για διάφορους λόγους η υπέρπτυση. Νομίζω ότι τα συστήματα μέχρι τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με κοινό τρόπο από τις αρχές ελέγχου και εποπτείας και των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις ε, για την ένταξη των μικρών και μεσαίων τηλεκατευθυνωμένων μηχανισμών ε, στον, ε, στους ουρανούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται λοιπόν οι μελλοντικοί κανόνες να είναι συμβατοί με τις διεθνείς συμβάσεις, να την χάνουν αμοιβαίας αναγνώρισης και ε, κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης της Επιτροπής Τραν για την επικοδομητική τους έκθεση, τη συνεργασία τους και τους συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, ιδιαίτερα τον Πάτρικ Κάσιντι από την ομάδα των συντηρητικών που με βοήθησε ιδιαίτερος. Νομίζω ότι όλοι είδαμε τις ευκαιρίες τις οποίες η αναδυόμενη αυτή αγορά παρουσιάζει στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, όπως επίσης και της κάλυψης των συμφερόντων των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το νέο εξαιρετικά τολμηρό και χρήσιμο βήμα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Σας Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, τα drones είναι μια τεχνολογία που ήδη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα πράγματα και δημιούργησε νέες ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες, για νέες εφαρμογές. Τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα μπορούν να επιτελέσουν αποστολές που ούτε μπορούσαμε να διανοηθούμε ούτε και ήταν οικονομικά εφικτές με επανδρομένα οχήματα ε, ελέγχους για λόγους ε, ασφάλειας, ε, παρατήρηση, αξιολόγηση των φυσικών καταστροφών, και ούτω καθεξής. Για την πολιτική χρήση αναπτύσσονται ραγδαία νέες τεχνολογίες και έτσι αυτός ο κλάδος μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. να αναγνωρίζουν το δυναμικό των νέων τεχνολογιών, όμως ταυτόχρονα εκφράζονται και ανησυχίες για τις αποστολές των drones και εξού και μια πρόκληση να θεσπίσουμε κανόνες που θα είναι εξισορροπημένοι, δηλαδή να προωθήσουμε τις νέες τεχνολογίες, όμως ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τους πολίτες μας για να γνωρίζουν ότι μόνο ευρωπαϊκοί κανόνες θα αποτελούσαν μια ισχυρή βάση για να προσελκύσουμε επενδύσεις αλλά και να διευκολύνουμε τη χρήση των τεχνολογιών ενώ ταυτόχρονα ε, προστατεύουμε κατά το δεν την, τους πολίτες μας και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει θερμά την υποστήριξη για την έκθεση Φώστερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα στην εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και τις προσπάθειες ούτω ώστε να πηχούνται οι απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων μέσα σε αυτήν τόσο περιεκτική έκθεση. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκκληση της έκθεσης για ξεκάθαρους, εναρμονισμένους ρυθμιστικούς κανόνες ε, καταργώντας το όριο των 150 κιλών ε, που ισχύει τώρα ε, και που τηρούν τις, ε, οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει όριο βάρους. Όμως, προσοχή, δεν χρειάζεται βαριά νομοθετική ρύθμιση για όλα τα οχήματα. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή επιχειρησιακή προσέγγιση ώστε να είναι αναλογικοί οι κανόνες σε σχέση με το ποσοστό, το επίπεδο κινδύνου κάθε επιχείρησης. Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Πολιτικής ε, Αεροπορίας ε, και το Γιάρους, η Ένωση των Εθνικών Αριθμιστικών Αρχών, συνεργάζονται και με εμπειρογνώμονες από τις ΕΙΠΑ, από τον Καναδά, από την Ιαπωνία, ούτως ώστε να καταλήξουν σε κανόνες οι οποίοι θα συναδούν με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς ή της πολιτικής αεροπορίας, ούτως ώστε κάθε χρήστης drone να συνειδητοποιεί ε, μέσω ενημερωτικών φυλαδίων τους κινδύνους και τους κανόνες που ισχύουν θα πρέπει ο πιλότος ε, να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ε, και για μεγαλύτερες αποστάσεις θα πρέπει να ξέρουμε ότι μειώνεται ε, σε μεγάλο βαθμό το κόστος της επιχείρησης. Βλέπουμε εκεί ευκαιρίες για καινοτόμες επιχειρήσεις και φυσικά πρέπει να βρούμε επενδύσεις για την έρευνα και την τεχνολογία γιατί υπάρχουν κενά στην τεχνολογία. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη επιχειρήσεων drones όμως ρόλο κλειδί παίζει και η στάση των πολιτών. Οπότε η εφαρμογή ε, κανονισμών για την ασφάλεια και για την προστασία των ατομικών δεδομένων έχει ιδιαίτερη σημασία για να καλύψουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Η περιβαλλοντική προστασία, η ασφάλεια και η απόδοση ευθυνών συγκεκριμένα στον κλάδο των drones είναι άλλα ζητήματα που πρέπει να καλύψουμε. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι καλωσορίζουμε την έκθεση για τα drones σε μεγάλο βαθμό θα συμβάλλει στη μελλοντική θέσπιση κανόνων ασφάλειας καθώς και στις προϊούσες εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσμιση ενός ξεκάθαρου νομοθετικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα ντρόνς ε, και ταχύτατα στο άμεσο μέλλον ε, θα προχωρήσουμε ε, με την υποβολή πρόταση. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα την κυρία Πόστα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι ο και περισσότερο στην κοινωνία μας βλέπουμε και για την πολιτική αεροπορία και για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ε, ε, να ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται τα drones για την μαζική παρακολούθηση και ξέρουμε πόσο εύκολο είναι κάποιος σήμερα να αγοράσει ένα drone. Δεν υπάρχει όμως κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε αυτό και πρέπει να αντισταθούμε στα εμπορικά συμφέροντα. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιους κινδυνούς επισηρεί η εμπορική χρήση των εναέριων μη επανδρομένων εχημάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει θα καταθέσει μια νομοθετική πρόταση. Όλοι πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς όμως. Θα πρέπει να δούμε πώς οι υπηρεσίες, εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν αυτά τα εναέρια οχήματα, ώστε να μην παραβιάζονται βασικές προσωπικές ελευθερίες. Σας ευχαριστούμε. Τώρα προχωρούμε στο ΕΛΚ. Μιζελιέ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θέλω βεβαίως να ευχαριστώ την κυρία Φόρστερ για την έκθεση που κατάρτισε και παρουσίασε, όπως και τις άλλες πολιτικές ομάδες για την καλή του δουλειά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθεσία ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο των μεγάλων διεθνών ανταγωνιστών όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Μόνο κάποιες αρχές νομοθετικής παρέμβασης υπάρχουν σε κράτη-μέλη. Εμείς βέβαια στην Ευρώπη έχουμε τα περισσότερα δρόμους, πάνω από το 5% των μη επανατρεμένων αεροσκαφών, με 4 δις ε, σε κύκλο εργασιών και πάρα πολλέ χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να έχουμε ηγετική θέση λοιπόν και στο μέλλον θα πρέπει να ορίσουμε τους κανόνες που θα επιβληθούν σε παγκόσμιο επίπεδο με τις τεχνολογικές προδιαγραφές και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιβάλλουμε και τα δικά μας οράνματα, όπως συνέβη και με το GSM για τα κινητά τηλέφωνα. Πρέπει η Πρόεδρος, κύριε Μιζελιέ, κύριε Μιζελιέ, ήρεμα. Πρέπει να εγγυηθούμε λοιπόν απόλυτη η προστασία του πληθυσμού και ομαλή λειτουργία των ε, επιχειρήσεων με πολλές χιλιάδες ε, μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κανένα ατύχημα με νεκρό. Πρέπει να προστατεύεται η προσωπική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα. Με το να μας όμως τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών είναι σαν να βγάζαμε τον ε, φακό από μια φωτογραφική μηχανή πρέπει να, να προβλέψουμε, να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις και νομίζω ότι θα είμαστε κερδισμένοι. Ευχαριστώ 1,5 λεπτό έχουμε ρεστών και Δημοκρατών, ο κύριος Τσέμκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερο στην εξή τοποθέτηση. Έχουμε καθημερινά όλο και περισσότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται. Πετάνε πάνω από το κεφάλι μας στην Ευρώπη. Πολύ καλό αυτό μεν. Ταυτόχρονα σημαίνει σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία. Ότι τα drones θα τα έχουμε κοντά μας από εδώ και μπρος. Άρα χρειάζεται νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν νομοθεσία που ε, διέπει την χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η δική μου πολιτική ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκρατές, ε, θεωρούν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση εδώ, γιατί πρόκειται για ένα χώρο όπου πρέπει να υπάρχει ρύθμιση πανευρωπαϊκή. Η πολιτική χρήση των μη επαδρομένων αεροσκαφών δεν μπορεί να, περιοριστεί στα εθνικά σύνορα και θέλω ιδιαίτερος να σημειώσω ότι πρέπει να, να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και κυκλοφορία αυτών των drones και επίσης ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Η έκθεση της κυρίας Φώστερ είναι ένα πολύ αξιόλογο, ενδιαφέρον και πολύτυπο έγγραφο και υπογραμμίζει ακριβώς αυτές τις δύο πτυχές ως όφιλε την ασφάλεια δηλαδή και την προστασία του ιδιωτικού βίου τις παρουσιάζει πολύ ξεκάθαρα η έκθεση της κυρίας Φώστερ, την οποία θα υποστηρίξει η ομάδα μας. Ευχαριστώ κύριο οι ε, συντηρητικοί μεταρρυθμιστές. Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε ακόμη ένα φαινόμενο όπου η τεχνολογία προχωράει πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσει και η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προσδιοριστούν οι όροι της χρήση των drones, να εξασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Η κυρία Φώστερ έχει κάνει μια πολύ καλή ισορροπημένη πρόταση. Την έχει καταθέσει για διάλογο στο Κοινοβούλιο. Η έκθεση φυσικά δεν σκοπεύει να προδικάσει μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και εγώ θέλω να σημειώσω ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν υπερβολικοί περιορισμοί στη χρήση των drones, ειδικά αυτών που έχουν χρήση ψυχαγωγική ή άλλων. Δηλαδή δεν πρέπει να περιορίσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη στις μελλοντικές Ευχαριστώ, Φαν Μίντελμπουργκ. Eh, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φώστερ για μια εξαιρετική δουλειά. χρησιμοποιώντας το λογοπαίγνιο στην αγγλική well done, well drawn. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να νομοθετήσει το τεχύτερο δυνατόν για την χρήση των συγκεκριμένων μηχανισμών. θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε θέματα υπευθυνοποίησης των χρηστών. Πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για την ασφάλεια της χρήσης των τηλεχειριζομένων αυτών υπταμένων μέσων. Θα πρέπει επίσης τα μέσα αυτά να είναι ανοιχνεύσιμα κάτω από οιασδήποτε συνθήκες. Μία από τις προτάσεις οι οποίες γίνονται είναι να υπάρχει μια ηλεκτρονική σήμανση κάθε τέτοιου μηχανισμού. Θα μπορούσε να ενταχθεί στο πακέτο για τις αερομεταφορές στον μήνα Δεκέμβριο και ελπίζω ότι και με την επόμενη Προεδρία, την Ολλανδική, θα μπορέσουμε εμείς να διασφαλίσουμε την βιομηχανία των τηλεκατευθυνωμένων. Ο κύριος Κλέτς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Μπούλτς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φώστερ. Ε, επέδειξε πνεύμα συνεργασίας για την προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Είναι αποστολή και ευθύνη της Ένωσης να αναπτύξει νομοθετικές ρυθμίσεις για τον τομέα ε, των τηλεκατευθυνωμένων αεροσκαφών, να γίνουν οι σωστές διακρίσεις για την ερασιτεχνική χρήση και την επαγγελματική χρήση ε, των ε, υπταμένων αυτών μέσων. Είναι μια βιομηχανία που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, πράσινες θέσεις απασχόλησης και ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες όπως και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν κέντρα ανάπτυξης και να υπάρξει συνεργασία και με τους χρήστες αυτών των μέσων. Η ανάπτυξη της καινοτομίας θα διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και θα διασφαλίσουμε επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, νομίζω ότι εδώ τίθεται το θέμα συγκεκριμένα της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας. Λούντγκρεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αυξάνεται η δραστηριότητα με τα ντρόνους, εκεί είναι πραγματικά μεγάλο το δυναμικό. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες για την νέα αγορά, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική συμβολή χάρη στα ντρόνους στην οικονομία. Υπάρχει σκεπτικισμός σε σχέση με το αν χρειάζονται τα ντρόνους και ε, θεωρούν κάποιοι ότι ε, παραδείγματο χάρη χρησιμοποιούνται τα drones από τρελούς ε, παρανοϊκούς ε, που θέλουν να παρακολουθήσουν τους άλλους. Όμως δεν αναγνωρίζουν ότι μπορούμε παραδείγματο χάρη με χάρη στα οχήματα, εναέρια οχήματα να μετακινούμαστε πλέον τόσο πολύ εύκολα. Μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή ότι μπορεί η νέα τεχνολογία να αναπτυχθεί και μπορούμε να ρυθμίσουμε πολλά προβλήματα που τώρα δημιουργούνται. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε Ποιε είναι οι πρακτικέ δυνατότητε που προσφέρουν αυτά τα οχήματα και η βιομηχανία μπορού, μπορεί να δημιουργήσει πολλέ νέε ευκαιρίε, όμω αυτό προϋποθέτει ξαναλέω ξεκάθαρου κανόνε, ε, διότι προ το παρόν επειδή υπάρχει αυτή η άγνοια δεν τολμάει καμία εταιρεία να επενδύσει πολλά κονδύλια διότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι κανόνε. Η ακαιρεότητα είναι επίση ε, των ατομικών δεδομένων είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα διότι μπορεί να, εκεί που καθόμαστε και πίνουμε καφέ να ε, έρχεται από πάνω μας ένα ντρόουν και να μας παρακολουθεί. Θα πρέπει λοιπόν να μην παραβιάζονται βασικές ελευθερίες, να διατηρείται η κυριότητα των ατομικών δεδομένων, αλλά να συνειδητοποιήσουμε και ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες. Ευχαριστούμε κύριος, ε, η κυρία Αγνοτού. Κυρία Φώστερ, είναι πολύ καλή η έκθεσή σας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που δεν προσπαθείτε να προτείνετε τη ρύθμιση στρατιωτικών ενέργειων ε, οχημάτων. Ε, συμφωνώ επίσης με τις ανησυχίες σας, ε, διότι θέλετε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ένα ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε σχέση με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, παραδείγματο χάρη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί θα πρέπει να συζητήσουν τόσο ώστε να είναι ισόρροπη η νομοθεσία και να μας επιτρέπει ενώ προστασία τη ατομική ζωή ε, και προστασία των πολιτών, ναι, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούμε τι νέε τεχνολογίε. Όπω είπα και στην Επιτροπή, είναι απαραίτητο οι ευρωπαϊκέ και οι Εθνικέ αρμόδιε αρχέ να διατηρήσουν ένα περιθώριο ελιγμών, ώστε να αδειοδοτούν ή να απαγορεύουν τη χρήση των ντρόουν σε ε, προστατευόμενε ζώνε. Ε, επικροτώ την παράγραφο 42, όπου ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με Λοιπόν, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και στους μπλεκόμενους φορείς από τις ΕΠΑ. Δεν βλέπω τον κύριο Γκόλνες, οπότε θα δώσουμε τώρα το λόγο, λέει η Πρόεδρος, στον κύριο Μαρινέσκου. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Δεν θέλετε. Κύριε Μαρινέσκου, δεν θέλετε να λάβετε το λόγο. Μα δεν είναι εδώ ο κύριος Γκόλνης. Α, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν το είχα καταλάβει. Και σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, υπήρξε εποχή που το ίντερνετ ανήκε στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας, ενώ τώρα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της οικονομίας και βέβαια φέρνει πολλές άλλες εξελίξεις θετικές και αρνητικές της ε, κοινωνίας μας. Και γι' αυτό χρειάστηκε η ρύθμισή του, όπως και στα ε, μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πριν από μερικά χρόνια ακόμα ήταν κάτι πολύ σπάνιο αλλά και ακριβό. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησαν ορισμένες δειλές ε, δοκιμές στον χώρο της πολιτικής χρήσης, ενώ τώρα πια είναι κάτι το τετριμένο. Χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους, συμβάλλουν στην οικονομία ε, και βέβαια μπορεί να, να δημιουργήσουν και πολλά προβλήματα εάν ε, κινδυνέψει η ασφάλεια των εναέριων μεταφορών. Όλοι χρειαζόμαστε τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Ε, είναι ένα ζήτημα πια που έχει μετατραπεί σε ε, ζήτημα μαζικής χρήσης. Έχουμε ε, ανάγκη λοιπόν να εισαγάγουμε τη σχετική νομοθεσία. Η έκθεση κυρία Φώστερ είναι πολύ καλή, καλύπτει διάφορα θέματα, αποτελεί μια καλή βάση για νομοθεσία στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει μια ιδιαίτερη προσέγγιση καθώς είναι και ιδιαίτερο το ζήτημα. Μιλούμε για ένα αεροσκάφο σε τελευταία ανάλυση, άρα πρέπει να υπάρξει ζήτημα ε, επαλήθευσης και των όρων κατασκευής και της πιστοποίησης, όλα τα τεχνολογικά δηλαδή στοιχεία του αεροσκάφους, η διάκριση μεταξύ της πολιτικής και στρατηγικής χρήσης και της ψυχαγωγίας ε, και στον τομέα αυτό δεν έχουμε περιθώριο για περισσότερες καθυστερήσεις. Ευχαριστώ το Παρτέλα ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η χρήση των ε, τηλεκατευθυνόμενων μη επιδρομένων ενέργειων ε, ε, οχημάτων ανήκει στον χώρο του μέλλοντος. Έχουμε πολλά που έχουν αναπτυχθεί για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και πολλά ακόμη που αναπτύσσονται καθημερινά για πολιτικές χρήσεις. Ξεκίνησαν με τη γεωργία, στη διάσωση, σε άλλες δράσεις. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα εύχριστα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη που καθοδηγεί ο άνθρωπος και, και μπορεί έτσι να έχει πρόσβαση σε πολύ απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο για τα τηλεκατευθυνόμενα εναέρια οχήματα με τήρηση των όρων της ΙΚΑΟ και Ξέρουμε βεβαίως ότι θα, είναι, ε, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις στον χώρο αυτόν, άρα πρέπει να προβλέψουμε και την πιστοποίηση για τους τεχνικούς όρους κατασκευής, αλλά και καθοδήγησης ε, από τους λεγόμενους πιλότους αυτών των σκαφών. Η κυρία Φανβάζοϊτ. Θα υπερψηφίσω την έκθεση της Τζάκη Φώστερ. Έχει βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη μία πλευρά στην υποστήριξη σε μία αναδυόμενη βιομηχανία και από την άλλη στην προσπάθεια για διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα της υπερβολικής διακανονιστικής δραστηριότητας και έτσι πνίγουμε τον πολίτη μέσα σε ρυθμίσεις και κανονισμούς που θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια τη βιομηχανία. Αντίθετα στην έκθεσή της η κυρία Φώστερ ισορροπεί τον σεβασμό της ιδιωτικότητας, ε, τη νέα τεχνολογία, το σεβασμό του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παρά να παρακολουθήσει τις προτάσεις αυτές. Ο κύριος Ρικέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. κάποτε ήταν μόνο σε στρατιωτική χρήση ε, ε, τα drones, τώρα χρησιμοποιούνται γενικότερα ακόμα και, στην, ε, και στο γύρισμα κινηματογραφικών ταινιών. Η έκθεση Foster ορίζει σωστά τις λύσεις για τα ειδικά προβλήματα που δημιουργεί η χρήση των τηλεκατευθυνωμένων συστημάτων πρέπει να υπάρξει εναρμονισμός των προβλέψεων λειτουργίας του στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι θετικό για μια βιομηχανία αναπτυσσόμενη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως για κάποιες από τις πλευρές που υπογραμμίζονται όπως η προστασία της ιδιωτικότητας, αντιμετώπιση κινδύνων, διάκριση επαγγελματικής από ερασιτεχνική χρήση, ε, διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να βρούμε και τα μέσα να προασπίσουμε την βιομηχανία μας αυτή από τις επιθέσεις του υπόλοιπου κόσμου. Ναι λοιπόν στην έκθεση Φώστερ. Σέιμουρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ε, προσπάθεια διακανονισμού λέει η κυρία Φώστερ. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες ε, σύμφωνα με την παράγραφο 22 προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφαιρέσουμε την δυνατότητα των εθνικών αρχών να ελέγχουν την δραστηριότητα αυτή και να μην υπάρχει και δυνατότητα ε, ε, περαιτέρω ερμηνείας του τι αποτελεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η εθνική δραστηριότητα. Κυρία Σέιμορ, να μιλάτε λίγο πιο αργά γιατί δεν σας παρακολουθούμε, λέει η Πρόεδρος. Ε, συγγνώμη Πρόεδρε, λέει η κυρία Σέιμορ και στην παράγραφο 48 ζητείται ένας μηχανισμός ε, παρατήρησης και αναφορών. Ε, πώς ακριβώς ε, το εννοείτε. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων, του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι εναντίον κάποιων πολύ περιοριστικών διατάξεων και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα λόγω της έλλειψης διαφάνειας στη δραστηριότητα αυτή την τόσο πολλά υποσχόμενη. Θα καταψηφίσω την πρόταση. Ρεβόνταλόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να χαιρετήσω την προσπάθεια της κυρίας Φώστερ και των σκιωδών. Αποδεχόμενη την έκθεση αυτή σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοπορούμε για την δημιουργία ενός πλαισίου για την λειτουργία των τηλεκατευθυνωμένων βασικό για την λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί τις προτάσεις της κυρίας Φώστα. Πρέπει να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη προσοχή σε σχέση με τον έλεγχο των drones όπως επίσης και με το θέμα του καθορισμού απαγόρευσης υπέρπτυσης συγκεκριμένων περιοχών. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μελλοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την διάκριση ανάμεσα στην ερασιτεχνική και εμπορική χρήση. Με την πρόταση σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα στον τομέα των αεροπορικών για την ανάπτυξή του και ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήγατε πολύ γρήγορα λέει η Πρόεδρος, περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ένα λεπτό η κυρία Μοντέιρο, αν ακούσαμε καλά. Ευχαριστώ. Η χρήση των μη επανδρομένων αερίων οχημάτων στην πολιτική αεροπορία σχετίζεται με την ανάδυση νέων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Είναι ένας κλάδος όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό ρόλο, όμως ταυτόχρονα όπως ακούμε στη συζήτηση να έχουμε μια αναλογική και ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση. Δεν πρέπει να παρεμποδίσουμε το δυναμικό αυτής της αναδυόμενης αγορά. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να γίνει σεβαστή η προστασία τη ιδιωτική ζωή των ατομικών δεδομένων και, τη ε, και της ασφάλειας των πολιτών. Είναι περίπλοκο το ζήτημα και χρειαζόμαστε νομοθετική ρύθμιση. Αυτές ε, οι επιχειρήσεις ε, νέων τεχνολογιών μόνο έτσι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην έρευνα, στην καινοτομία και στην παροχή νέων υπηρεσιών. Υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να υπερβούμε σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε πολλά κράτη κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε ως εκ τούτου ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτω ώστε να μην δημιουργηθεί περιττή επιβάρυνση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Εγώ θα υπερψηφίσω αυτή την έκθεση. Ο κ. Φρουντσούλικα. Dear colleagues, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι όντως ε, η ώρα να εξασφαλιστεί ένα εναρμονισμένο και ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα μη επανδρομένα τηλεκατευθυνόμενα εναέρια οχήματα και εν ώψη της ε, δέσμης μέτρων που αναμένεται να κατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αεροπορία. Και αυτά σύμφωνα με την διακήρυξη της Ρήγας, με εξασφάλιση της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ιδιωτικού βίου δηλαδή και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να προωθηθεί η χρήση των μέσων και της τεχνολογίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα 150 κιλά ως όριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι νομίζω ένα όριο που θα πρέπει να ορίσουμε. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στην εποχή της τεχνολογίας θα μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα σε σχέση με την έρευνα και τη διάσωση, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, τη δημοσιογραφία, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες αναψυχής. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει άμεσα μέτρα, έτσι ώστε τα τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπού εξυπηρέτηση των ίδιων των ανθρώπων. παράλληλα η ευρωπαϊκή επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα καθώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι εξ ορισμού μια μορφή τεχνολογία διπλή χρήση και απαιτείται έτσι η επιβολή περιοριστικών και αυστηρών κανόνων προκειμένου να υπάρχει προστασία τη ιδιωτική ζωή και των προσωπικών δεδομένων. παράλληλα τα συστήματα αυτά μπορούν είτε σκόπιμα είτε όχι να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν ανθρώπου και υποδομές εφιστώ λοιπόν την προσοχή της επιτροπής για τα τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη και ζητώ να υπάρξει συγκεκριμένη παρέμβαση νομοθετική. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε θέλω να ευχαριστήσω, να συγχαρώ μάλλον την κυρία Φώστερ για τις απαιτούμενες προτάσεις ρυθμίσεων για τα μη επανδρομένα αυτά μέσα. Το χρειάζεται ο τομέας σε έναν τομέα όπου ο διεθνής ανταγωνισμός είναι παρόν. Απαιτείται και οι κατασκευαστές και οι πολίτες να έχουν συγκεκριμένα πεδία αναφοράς για την προστασία τους και την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την δυνατότητα συντονισμού με τις υπόλοιπες αεροπορικές δραστηριότητες κάνοντας τη διάκριση ανάμεσα στην επαγγελματική ε, και ερασιτεχνική χρήση και να αποφύγουμε κατεχρήσεις στον τομέα της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν τον κίνδυνο τον οποίο μπορεί να παρουσιάζουν οι τεχνολογίες διτής χρήσης σε μια νέα ευκαιρία και στη δημιουργία θέσεων ποιοτικών μάλιστα απασχόλησης. Ευχαριστώ. Σούλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε τα συστήματα μη επανδρομένων μερίων οχημάτων όταν δεν ε, ε, καθοδηγούνται από κατάλληλα καταρτισμένους ε, ανθρώπους συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, για την, την προστασία των ατομικών μας δεδομένων, για την υγεία των ζώων. Χρειαζόμαστε αυστηρότατη ρύθμιση και ψηλότατο πρότυπα ακόμη και για τις κατασκευαστικές ετάλια και προστασία της ιδιωτικής ζωής έχουν ζωτική σημασία όπως αναφέρεται στην έκθεση και τα πρόσφατα σκάνδαλα με τη χρήση των drones μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθήσουμε και την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων με κατάλληλο τρόπο. Χρειάζονται επίσης πηγές χρηματοδότησης ε, και είναι, επικροτούμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσέλκυση επενδύσεων. Υπάρχει ένα σοβαρό κενό στην νομοθετική ρύθμιση και γι' αυτό χρειαζόμαστε συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τα θέματα ασφαλείας προστασία του περιβάλλοντος και προστασίας προστασία ιδιωτικής ζωής. Ε, κύριε Άντερσον, καλημέρα σε όλους. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω την συζήτηση που γίνεται και επίσης τον τρόπο με τον οποίο εκπονήθηκε η έκθεση, ε, διότι έτσι αποφεύγουμε από τους, ε, τα, τα κακοπροαίρετα σχόλια των Βρετανών συναδέλφων που κάθονται στην απέναντι πλευρά του ε, ε, ε, ε, είναι ξεκάθαρο ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τι επιδιορθώσει για την επιτήρηση στον κατασκευαστικό τομέα. Ε, υπάρχουν επικίνδυνες επιχειρήσεις για τους ανθρώπους που μπορούν κάλλιστα να επιτελεστούν από μια επανδρομένη ενέργεια οχήματα. Όμως υπάρχουν και σοβαρά ατυχήματα που έχουν ήδη συμβεί στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Γι' αυτό είναι απογοητευτικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να νομοθετήσει εξίσου αυστηρά και την χρήση για για αναψυχή των drones. Ε, φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Ε, Όμω ε, στον τομέα τη χοντρική και λιανικής θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την προστασία τη ασφάλεια και των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστούμε. Ε, ολοκληρώνοντα τώρα το CATSDI. Ο κύριος Γιάκοφτη, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κύριε επιτροπα. να εκφράσω την υποστήριξή μου την έκθεση της κυρίας Φώστερ, η οποία αναφέρεται σε οχήματα των οποίων η αγορά έχει τεράστιο δυναμικό ανέπτυξης και χρήσης. Θα ήθελα ιδιαίτερα δε να σας επισημάνω τα εξής. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό και κατάχρησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών, άπαξ και ενταχθούν στην καθημερινή μας ζωή και αρχίσουν να πετάνε κατά χιλιάδες πάνω από το κεφάλι μας. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι πώς θα τα εντοπίζουμε, πώς θα αναγνωρίζεται, πώς θα ταυτοποιείται ο χρήστης τους ή ο κύριος τους, πώς θα ελέγχεται ο τρόπος πτήσης και ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η υπερσυνοριακή χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών όπου εφόσον διασχίσει ένα ε, μια συνοριακή γραμμή των drone, ε, τίθενται ζητήματα και ασφάλειας. Η κυρία Μπούλτς, πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ. την επικοδομητική συζήτηση. Η βιομηχανία των μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη, για την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, για τα επαγγελματική χρήση οχήματα, ενέργεια οχήματα πρωτοπόρος. Δεν θέλουμε να παραμείνει πρωτοπόρος. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε ένα συγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, του τρόπου λειτουργίας της ε, και, και πρόθεση της ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για μια αγορά που προχωρά ταχύτατα, εξελίσσεται ταχύτατα. Θέλουμε μια ταχεία και ολιστική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Είπαμε ότι στην δέση μέτρων για την αεροπορία θα καλύψουμε ζητήματα της εκθέσεως και δραστηριότητες της ΕΑΣΑ και της ΓΙΑΡΟΥΣ. Η τεχνολογία και η παραγωγικότητα της βιομηχανίας ε, πρέπει να εξισορροπηθούν με την ασφάλεια, την ε, προστασία του ιδιωτικού βίου, την αποφυγή της χορύπανσης και βέβαια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χρήστη του drone. Πρέπει να ε, λάβουμε μια προσέγγιση ισορροπημένη ώστε να προβλέψουμε τις εξελίξεις αγοράς και την εκδήλωση των διαφόρων πτυχών. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την κυρία Φώστερ και όλους τους ευρωβουλευτές που έλαβαν μέρος ε, στην κατάρτιση της έκθεσης και προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία στο θέμα αυτό. Η κυρία Φώστερ παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ε, επικοδομητικές τους παρατηρήσεις. Να κάνω ορισμένε διευκρινήσεις. Καταρχάς για την ε, εμπιστευτικότητα, ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Γνωρίζουμε ότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν ισχυρές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν. Νομίζω λοιπόν ότι από από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για τα λεγόμενα baby drones, τα πολύ μικρά αυτά μέσα. Ε, βασικός στόχος της έκθεσης αυτής είναι ο μεσαίος τομέας, όχι αυτά τα μικρά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και από εμπορικές επιχειρήσεις και μπορεί να προκαλέσουν ε, ζημίες και δεν μιλάμε για τις ε, μεγάλες μηχανές που καλύπτονται ήδη από τις ρυθμίσεις των αερομεταφορών. Σχετικά τώρα με την προστασία των ε, εγκαταστάσεων όπως οι πυρηνικές μονάδες, τα αεροδρόμια κτλ. Εδώ τίθεται το θέμα του λεγόμενου geofencing, δηλαδή της προστασίας και της απαγόρευσης υπέρπτυσης. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε και για την συνάδελφο Αρνοτού. Το θέμα δεν αφορά τη στρατιωτική χρήση. Μιλάμε για την πολιτική χρήση στην παρούσα φάση. Και ένα τελευταίο σημείο, μια τελευταία παρατήρηση μετά από αυτά τα οποία είπε η κυρία Σίμουρ η οποία δεν κατανοεί πραγματικά τον τομέα των αερομεταφορών. Δεν κατανοεί ότι οι αερομεταφορές ελέγχονται από εθνική, επίσης ευρωπαϊκή και παγκόσμια ρυθμιστική θα έλεγα έλεγχο, εποπτεία. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από την παρατήρηση να πω ότι προσβλέπω ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζω να προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση το ταχύτερο δυνατόν οι κατασκευαστές, οι χρήστες και όσοι μίλησα θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή τη συζήτηση όπως και εμείς ε, σαν νομοθέτες. Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω να υποστηρίξετε όλοι στις, ε, στην ψηφοφορία στις 11.30. Πράγματι η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα.